Να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές. Η ψηφοφορία θα λάβει χώρα αύριο. Η επόμενη συνεδρίαση αύριο στις 8.30 ε, η ώρα το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι και μετά μέχρι τις 5. Η ημερήσια διάταξη έχει δημοσιευτεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και τους ήρμηνες. Καλό σας βράδυ.